Please can may to to Παρακαλώ καθίστε συναδελφοί, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας ε, τον Επίτροπο, τον κύριο Ερτέγκερ, τον οποίο και ευχαριστώ για την ε, παρουσία του εδώ σήμερα, για την ειδική αυτή συνάντηση της Επιτροπής μας και επίσης επειδή καταφέρουμε να διοργανώσουμε αυτή την ειδική σε. Και να συνεχίσω στα Ιταλικά. Έχουμε τρία μικρά σημεία να διεκπαιρέωσουμε. Καταρχάς, ε, συμφωνείτε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αν έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη όπως διατυπώνεται. Αλλιώς έρθει εγκεκριμένη. Κατά δεύτερον, για τη διερμηνία σήμερα το απόγευμα. Έχουμε γαλλικά, γερμανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Ελληνικά μπορείτε και να ακούσετε και να μιλήσετε. Come sapete, questo incontro è trasmesso in web streaming. Και τώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο αρμόδιο για την ψηφιακή οικονομία και την ψηφιακή κοινωνία, τον κύριο Γκουστάβ Ερτιγκερ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας καλωσορίζω εδώ σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που ε, επισκέπτεστε την δική μας επιτροπή Έγινε ψηφοφορία υπέρ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ε, είδαμε τότε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων και νομίζω ότι μπορούμε να διοργανώσουμε τη συζήτησή μα ω εξή. Θα έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα να κάνετε τα εισαγωγικά σα σχόλια. Μετά θα έχουμε μια, ένα πρώτο γύρο έρωτα απαντήσεων από του συναδέλφου και θα ακολουθήσει και μετά ένα δεύτερο γύρο με πιο συγκεκριμένε ερωτήσει. Επιτρέψτε μου όμω να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια για ε, κάποια ζητήματα που μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα. Ακούσαμε και στην ακρόαση ότι μιλήσατε και να σας υπενθυμίσω ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια διαφορετική σύνθεση. Τα θέματα ψηφιακής οικονομία είναι στην Γενική Διεύθυνση Econet και χαίρομαστε φυσικά που ε, αυτά εντάσσονται σε μια συνελική προσέγγιση από πλευρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που θα μας ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε από εσά ε, τι γίνεται με θέματα χρονοδιαγράμματος σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ε, οπτικοακουστική οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Λάβαμε και κάποιες υποδείξεις ότι το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2016. Μας απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάχθηκε υπέρ μια ταχεία αντιμετώπιση και διεκπαιρέωση του θέματο, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση στον τομέα αυτό. Και ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να αναφέρω, κάτι που και εμά μα απασχολεί πάρα πολύ, το θέμα της ε, Creative Europe, Δημιουργικής Ευρώπης. Ε, συζητήσαμε με τον αρμόδιο επίτροπο και του είπαμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται σε διάφορες ε, αρμοδιότητες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλαμε λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα το πώς συγκεκριμένα διαμορφώνεται αυτή η συνεργασία και πρόκειται να διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά και τα χρηματοοικονομικά μέσα, τους πόρους που χρειάζονται. Είμαι βέβαιη ότι όλοι έχουν ε, πολύ ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και το θέμα του copyright ε, των πνευματικών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας μαζί με την Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή, την Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων. Είναι σίγουρα λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και περιμένουμε διευκρινήσεις από πλευρά σας. Κάποια άλλα ζητήματα, το θέμα της πολιτιστικής ε, Πώ ε, πώς μπορούμε να το ψηφιοποιήσουμε το περιεχόμενο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ε, Ευρωπαίοι που το θέτουν διαρκώ το θέμα αυτό. και άλλο ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Γενική Διευθυνσή Connect. Όχι μόνο για, τα, για το πρακτηρητήριο, για τα οπτικοακουστικά, αλλά για τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται εδώ πέρα και τα, θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας ε, άποψη. Ένα άλλο ζήτημα. Είδα ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker τονίζει και ένα θέμα που άπτωται τον... Ε, Τη εκπαίδευση και του ICT σε ό,τι αφορά τη χρήση των δορυφόρων, σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Θα θέλαμε να ακούσουμε πιο πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά και τη συνεργασία στον κλάδο αυτό. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτάσει να μα καταθέσει προ την κατεύθυνση αυτή, θα περιστώ σε αυτά. Ήθελα απλά να σα αναφέρω κάποια ζητήματα, αλλά φυσικά και οι συνάδελφοι θα θέσουν τα ερωτήματά του. Αξιότιμη κύριε Πέτρο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και για τα όσα είπατε εισαγωγικά. Γνωρίζω πολύ καλά ότι για τα καθήκοντά μου στην Επιτροπή δεν είναι αρμόδια μόνο μία κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά περισσότερε από μία. Αφενός έχουμε την Επιτροπή Ήτρε, ε, έχουμε την Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων, τη δική σα, την Επιτροπή Εσωτερική αγορά και με ενδιαφέρει πολύ να συζητήσουμε τις πρωτοβουλίες που έχουμε σκοπό να αναλάβουμε στην Κομισιόν ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη σχέση μας μαζί σας και να μπορείτε να λαμβάνετε από την πλευρά μου μελέτες, στοιχεία που συλλέγουμε στην Κομισιόν ή που συλλέγονται κατ' εντολή της ε, Κομισιόν για να μπορείτε κι εσείς να εμβαθύνετε στα ζητήματα αυτά. Θέλουμε επίσης την εσωτερική, να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Η Ευρώπη ε, είναι μια κοινότητα αξιών, είναι μια νομισματική ένωση και είναι και μια εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχουν λοιπόν εθνικά σύνορα για υπηρεσίες, αγαθά, ε, τραπεζικές υπηρεσίες, αυτοκίνητα, κλωστή φαντουργία. Για όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχει ενιαία αγορά, αλλά όχι στην ψηφιακή ε, οικονομία. Εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν 28 κατακερματισμένες αγορές. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δούμε και πώς έχει αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα σε άλλες περιφέρειες του κόσμου, στη ΣΥΠΑ, στην Νότια Κορέα στην ε, Κίνα, πώς ε, με αυτόν τον τρόπο ε, αμβλήθηκαν τα προβλήματα, πώς με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η οικονομία, αναπτύχθηκε η οικονομία και το όραμά μας μπορεί να συνοψιστεί υπό τον τίτλο «Θέλουμε μια ψηφιακή ένωση». Τον Μάιο ο συνάδελφος Άνζιπ, σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους, θα παρουσιάσουμε τη στρατηγική μας για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Αυτό που μπορώ να σας πω από τώρα είναι ότι υπάρχουν τα εξής δομικά στοιχεία για το 2015-2016. Πρώτον, θα υπάρξει κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είμαστε αρκετά αισιόδεξοι ώστε να πιστεύουμε ότι στο Συμβούλιο σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα υπάρξει συμφωνία για τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έως το τέλος του 2015. Κάποια στιγμή έχει κολλήσει η συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν στο Συμβούλιο, αλλά πλέον ε, επιταχύνονται οι διαδικασίες και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταφέρουμε να τη θέσουμε σε ε, ε, ισχύ Δεύτερος πυλώνας είναι η αγορά τηλεπικοινωνιών. Μετά από ε, συνάντηση που είχαμε τους είμαι, με τους υπουργούς, είμαι αισιόδοξο ότι η Λετωνική Προεδρία, ακόμη και το Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, θα λάβει την εντολή για να ξεκινήσει την πραγματεύση με το Κοινοβούλιο. Αυτά που μας απασχολούν είναι ο ορισμός για την ε, ουδετερότητα στο διαδίκτυο, ο χρονικός άξονας, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή για την εφαρμογή του roaming και το ερώτημα της, ε, του συντονισμού και της εναρμόνισης των συχνοτήτων στην Ευρώπη, του φάσματος συχνοτήτων δηλαδή. Να πω επίσης ότι και σε αυτό το θέμα υπάρχουν καλές, ε, καλή, υπάρχει καλή προόδος στο Συμβούλιο και θα αποτελέσει, αν τελικά καταλήξει η συμφωνία, ένα πρώτο βήμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζουμε ότι και αυτό θα είναι δυνατό, θα καταστεί δυνατόν πριν από το 2015, το τέλος του 2015. Copyright. Αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Τα, πνευματικά δικαιώματα ξέρετε ότι ρυθμίζονται σε πάρα πολλές νομοθετικές πράξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν τη φιλοδοξία το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο φέτος να υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση για σύγχρονα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα. Οι μελέτες, οι νομικές αξιολογήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν συλλεχθεί. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ορισμένες συνεδριάσεις από την πλευρά μου με διάφορους εμπλικόμενους φορείς για να επεξεργαστούμε ορισμένες τελευταίες πτυχές και έχουμε καταλήξει πλέον σε μια ισορροπημένη στάση. Και αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι αυτός που δημιουργεί με το πνεύμα του, ο σενεριογράφος, ο σκηνοθέτης, ο συνθέτης, ο ίδιος ο μουσικός, ο δημοσιογράφος που συντάσσει ένα άρθρο σε εφημερίδα, και που πριν από τη σύνταξη αυτού του άρθρου κάνει την έρευνά του. Υπάρχουν οι εκδότες και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι προσδοκίες των χρηστών του δικτύου να έχουν πρόσβαση σε όσο περισσότερο περιεχόμενο γίνεται, εφόσον αυτό είναι ψηφιακά διαθέσιμο. δημόσιες βιβλιοθήκες ε, έχουν ε, δικαιώματα πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και ποια ακριβώς είναι η αξιοποίηση όλων αυτών των δικαιωμάτων. Αν δεν υπάρχουν δικαιώματα χρήσης, πνευματικά δικαιώματα δηλαδή, για την πνευματική ιδιοκτησία, αυτό θα οδηγήσει στο θάνατο της πνευματικής δημιουργίας. Θα πρέπει δηλαδή να περιοριστούμε στο Σέιξπιρ και σε διάφορους ε, μουσικούς που έχουν ε, γράψει τη μουσική τους μέχρι σήμερα. Γιατί δεν θα μπορεί κανείς πλέον να ζήσει από την πνευματική δημιουργία. Τον, το καλοκαίρι λοιπόν ή το φθινόπωρο θέλουμε να παρουσιάσουμε την ομοθετική μας πρόταση με στόχο στη βάση αυτή άρθρο προς άρθρο να συζητήσουμε μαζί σας και να καταλήξουμε σε αυτήν την ισορροπία που περιέγραψα. Θέλουμε παράλληλα να υπάρχουν μάλλον παράλληλα και εθνική, εθνικές νομοθετικές πράξεις. Στη Γερμανία για παράδειγμα υπάρχει αντίστοιχος νόμος αλλά φαίνεται ότι αυτές οι εθνικές διατάξεις μάλλον είναι άνευ αντικειμένου, διότι οι παγκόσμιοι παίκτες, η Google, η, το Facebook και άλλοι, δεν ε, σέβονται τις εθνικές διατάξεις. Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν θα μπορούσαμε και με βάση τους νόμους για την ανταγωνιστικότητα να επιβάλλουμε συγκεκριμένους κανόνες. Αναφερθήκατε στην ε, οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι είμαι πολύ φιλόδοξος στο θέμα αυτό και ξέρω ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Φέτος θα ε, υποβάλουμε σε αναθεώρηση τη συγκεκριμένη οδηγία. Και στόχος μου είναι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση αυτή εντός του 2015. Ε, ίσως να μην διατυπώσαμε αρκετά φιλόδοξα το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Δεν θέλουμε να τελειώσουμε το 2016, θέλουμε να τελειώσουμε το 2015, ώστε αμέσως μετά να σας ρωτήσω και να καταλήξουμε σε απόφαση για το αν θέλουμε να ε, προχωρήσουμε σε αναθεώρηση. Με βάση τις ε, τωρινές μου εκτιμήσεις ε, θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση της οδηγίας αυτές. Και στόχος μου είναι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 να υποβάλουμε μια αναθεωρημένη έκδοση της οδηγίας ώστε εντός του 2016 να γίνουν οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Δεν θέλω να χρονοτριβώ. Στόχος μου είναι στο τέλος του 2015 να έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένη απόφαση και αρχές του 2016 να υποβάλουμε συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης, την οποία και θα υποβάλουμε σε εσά για να ε, την συζητήσουμε. Για το θέμα των πολιτιστικών πόρων μας και της ψηφιοποίησης αυτών, της ε, μετατροπής τους δηλαδή ε, σε ψηφιακή μορφή, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και παρά τους δημοσιονομικούς ε, περιορισμούς θα προσπαθήσουμε. Ξέρετε ότι η ψηφιακή συνιστόσα το Connecting Europe μειώθηκε από τα 9 στα, 1, στο 1 δισεκατομμύριο. Παρ' όλα αυτά θα κάνω ό,τι μπορώ μέσω ε, επενδυτικών ταμείων του Connecting Europe και άλλων χρηματοδοτικών μέσων να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη, για τις τοπικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ψηφιοποίηση του της πολιτικής μας κληρονομιάς. Αναφερθήκατε και στο επενδυτικό πακέτο Juncker. Αυτόν τον καιρό προετοιμάζουμε δύο ε, πυλώνες. Και χαίρομαι πολύ που ο Juncker θεωρεί ότι οι ψηφιακές επενδύσεις είναι σημαντικές στο πλαίσιο αυτού του πακέτου. Ότι τα χρήματα δηλαδή από το πακέτο δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σιδηρόδρομους και δρόμους, αλλά και για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, με τις τοπικές αρχές, με την Επιτροπή των Περιφερειών, με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, για να συζητήσουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε, ώστε να επεκτείνουμε την ευρυζωνικότητα, τις οπτικές είναι ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και πώς μπορούμε όλο αυτό να το καταστήσουμε εφικτό οικονομικά. Δεύτερον, skills, δεξιότητες, εκπαίδευση. Κάθε χρόνο χρειαζόμαστε 150.000 ε, ειδικού ε, στην ε, τεχνολογία πληροφοριών Και αυτό αφορά τα κράτη-μέλη, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θέλω να συζητήσω με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπινους πόρους στο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολίτες που θα διαθέτουν ψηφιακά προσόντα. Και σκεφτόμαστε αυτόν τον καιρό πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα voucher για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για άνεργους, με ευρωπαϊκά κονδύλια, για να μπορούν οι άνθρωποι σε λαϊκά πανεπιστήμια, σε, τοπικά, σε τοπικές σχολές, να παρακολουθήσουν μαθήματα πληροφορικής, πώς θα μπορούσαμε να συγκριματοδοτήσουμε τέτοια έργα και να αξιοποιήσουμε στον βέλτιστο βαθμό αυτά τα βάουτσερ, αυτά τα κουπόνια, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να αποκτήσουν ψηφιακά προσόντα στον ελεύθερο χρόνο τους και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν ικανότητες που τις χρειάζονται είτε κάνουν τις αγορές στο διαδίκτυο, είτε ε, στο ίντερνετ των πραγμάτων. Χρειαζόμαστε να εκπαιδεύσουμε, να εξοπλίσουμε τον πληθυσμό μας με αυτά τα προσόντα, με αυτές τις δεξιότητες. Αυτά είχα να πω από την πλευρά μου. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήματα που θα έχετε και που αφορούν και το δικό σας έργο εδώ στην Επιτροπή. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξή. Έχουμε περίπου μία ώρα μέχρι τις 5 με τον Επίτροπο να τηρήσουμε την χρονολογική σειρά που ζητήθηκε ο λόγος και να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους. Bardzo dziękuję. komisarzu, dwie kwestie. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Καταρχάς, αναφέρατε την αναγκαιότητα να κοιτάξουμε, να ξανακοιτάξουμε την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Θα μπορούσατε να φανταστείτε επίσης να διευκολύνουμε περαιτέρω την οργάνωση των ε, διεθνών σπουδών με την χρήση ε, μοντέρνων τεχνολογιών. Πιστεύετε ότι η οδηγία αυτή θα έπρεπε να διευκολύνει την ε, συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων. Και μία δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε τι προτάσεις υπάρχουν στη συμφωνία TTIP για τα δικαιώματα δημιουργού, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση των ε, διαφορών πόρων, παραδείγματο χάρη των βιβλιοθηκών, των μουσείων κτλ. Ο κ. Λούερς έχει το λόγο. Έχουμε 13 ομιλητές, θα τους διαρρέσουμε σε δύο ομάδες. Για να πάρουν το λόγο πρώτα η μισή και μετά η υπόλοιπη μισή. Ευχαριστώ. Ε, καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Η εξή ερώτηση θα σα τεθεί τώρα. Η Κομισιόν σκέφτεται να καταργήσει geoblocking. Το σκέφτεστε. Αυτό θα δημιουργήσει σε καλύτερη χρηματοδότηση του δημιουργικού περιεχομένου ή και θα υπάρχει περισσότερο περιεχόμενο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάνετε το μπλοκάρισμα, δηλαδή με βάση την γεωγραφική θέση η ε, κυρία Τρίπολη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζίνγκερ. Τέσσερι ερωτήσει έχω να σα κάνω. Εγώ είμαι από αυτού του βουλευτέ που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την. νέα αναθεώρηση της οδηγίας για τα οπτοακουστικά μέσα. Θεωρώ ότι δεν είναι πλέον, ε, είναι παροχημένη και πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξαναυπάρχει, να ξαναυπάρξει ρύθμιση της πλατφόρμας. Συμφωνείτε. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω ποιος θα είναι ο ορισμός της ουδετερότητας του δικτύου. Ύστερα, μιλήσατε για την Google. Θα ήθελα να, μου πείτε πώς το φαντάζεστε την προσέγγιση και άλλο ένα περίπλοκο θέμα. Η χρηματοδότηση του Euronet. Πώς θέλετε να γίνει. Ε, Ευχαριστώ. Για κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποτέ δεν διευκρινίστηκε το εξή η σχέση και η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αντιπροέδρων και των επιτρόπων σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες επικαλύπτονται, όπως στη δική σας περίπτωση, ας πούμε, ή κάποιες αρμοδιότητες. Ας πούμε ότι είναι μια ερώτηση που ξεφεύγει λιγάκι από το σημερινό θέμα. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του copyright, στο οποίο αναφερθήκατε. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερο, περισσότερες ευκρινήσεις σε δύο θέματα. Καταρχάς, την οδηγία για τις ε, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Στο πρόγραμμα εργασίας μιλήσατε για αξιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς για σας. Σε τι συνίσταται έτσι, με πολύ συγκεκριμένους όρους. Και δεύτερον, τα επόμενα βήματα της Κομισιόν, ποια θα είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί αφορά κυρίως την Νότια Ευρώπη. Η Κομισιόν έχει σκεφτεί να διαφυλάξει και να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται ε, με τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, που είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση. Για το θέμα του copyright τώρα, με βάση τα όσα μας είπατε εσείς πριν και τις διακήρυξεις που έκανε ο αντιπρόεδρο πριν από λίγε μέρε, ε, βλέπω ότι η κατάσταση του copyright είναι πολύ διαφορετική από κράτο σε κράτο. και επομένω, είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί η ψηφιακή αγορά. Μπορείτε να μα επιβεβαιώσετε λοιπόν εσεί ότι η πρόταση θα περιλαμβάνει έναν ορισμό του copyright και θα προβαίνει σε μια εναρμόνιση τη διάρκεια του copyright σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ε, ευθύνες των ενδιάμεσων, των μεσαζόντων δηλαδή. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά βεβαίω τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει όμως ε, την, αυτό το πράγμα το επιβλέπει μία δικαστική αρχή και όσοι και επομένως ε, όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες online να είναι υπεύθυνοι. Εμείς έχουμε πολλά προβλήματα στην Ιταλία. Επίση, κάτι άλλο. Εσεί προηγουμένω μιλήσατε για το copyright και μιλούσατε με οικονομικού όρους. Πώς οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους εάν δεν ε, υπάρχει μια ανταμοιβή, αν δεν, έχουν, ε, δεν πληρώνονται για αυτό που κάνουν. Να σας ρωτήσω το εξή λοιπόν. Φυσικά όποιο εδώ παραβαίνει θα πρέπει να τιμωρείται. Πώ θα προστατεύσετε την ε, διανομή πολιτιστικού περιεχομένου. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια α, παραδείγματα α πούμε. Παραδείγματο χάρη ε, ο Walt Disney, ας πούμε, ο οποίο ποτέ δεν πλήρωσε πνευματικά δικαιώματα, ε, χρησιμοποίησε ας πούμε, τους μύθους ε, Grimm, αλλά τους, μεταπεί, τους μετασχημάτισε ας πούμε, σε κάτι καινούριο. Σας παρακαλώ, λέει Πρόεδρος. Από εδώ και πέρα θα ήθελα λίγο πιο συνοπτικές ερωτήσεις. Ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Έτιγκερ για τα λόγια που μας είπατε και την παρουσίαση που μας κάνατε. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε ότι ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης εξασφαλίζεται και μέσω της ε, online παρουσίασης περιεχομένου. Αν κοιτάξουμε την νομοθεσία κάποιων κρατών μελών, υπάρχει ας πούμε περίπτωση της Ισπανίας με ένα νόμο που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο πέρυσι, του 2014 δηλαδή. Είναι ένας νόμος για το copyright που είναι πολύ αμφιλεγόμενος στη χώρα μου και θα, ε, θα επέβαλε ας πούμε ε, για να προστατεύσει την χώρια βιομηχανία να επιβάλλει φόρους σε Google κτλ. Πώς θα εξασφαλίσετε τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης σε αυτή την προσπάθεια μεταρρύθμισης της, και μέσα από την προσπάθεια μεταρρύθμισης της οδηγίας που θα μας ε, υποβάλλατε. Λοιπόν, ο τελευταίος ομιλητής από τον πρώτο γύρο ομιλητών. Ευχαριστώ κύριε Έτιγκελ για το γεγονό ότι ήρθατε εδώ σήμερα και θέλετε, είστε διαθέσιμο να απαντήσετε στα ερωτήματά μα. Για μένα υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα. Ορισμένα αναφέρθηκαν ή Θα ήθελα να ε, εμπαθύνουμε λίγο στο, ε, στο θέμα του Single European Title. Θέλουμε δηλαδή εδαφική προσέγγιση, εδαφική εμπορία περιεχομένου ή θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκές άδειες χρήσης, ε, θα πρέπει να, ίσως να θεσπιστούν ε, και τέτοια μέτρα. Δεύτερον, ιδιαίτερα όσον αφορά το copyright, χρειάζεται να υπάρχει απλούστευση της νομοθεσίας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, κάτι τέτοιο θέλετε να το κάνετε με οδηγία ή με κανονισμό. Δηλαδή με άλλα λόγια, θέλετε να το κάνουμε όπως το κάναμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλετε να ε, ορίσουμε κάποιες βασικές αρχές που θα εξειδικευτούν στα ε, κράτη-μέλη ή μια διαφορετική προσέγγιση θέλετε να υιοθετήσετε για το TTIP. Τι γίνεται με τον ορισμό των ε, οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Θα ε, εμπέσει στην κατηγορία της ε, ψηφιακής εξαίρεσης. Τα, τα οπτικοακουστικά μέσα θα θεωρηθούν ως τμήμα της πολιτικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Θα εμπέσουν δηλαδή στο TTIP ή θα εξαιρεθούν από αυτό. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ήθελα να σας ξαναπώ ότι και για την εκπαίδευση, για τις δεξιότητες, το θέμα δεν είναι μόνο να εκπαιδεύσουμε και να παράσουμε δεξιότητες στους μαθητές, αλλά και στους δασκάλους μας. Γιατί πολλές φορές έχουμε την ε, κατάσταση κατά την οποία οι μαθητές ε, έχουν περισσότερες ικανότητες και γνώσεις ε, περίπληροφορικές από τους, από τους καθηγητές τους. Από αυτή την άποψη θα είχε νόημα να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και στους δασκάλους. Και κάτι που αναφέρθηκε και ανέφερε η κυρία Τρούπελ. Μειώθηκαν πράγματι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα κονδύλια από το Connecting Europe. Όμως είπατε κι εσείς ότι θα αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του Euronews, του Europeana. Πρόκειται για ένα σύστημα που δημιουργήθηκε ακριβώς για να μεταδίδονται ευρωπαϊκού χαρακτήρα ειδήσει, για να ε, γίνονται προσβάσιμες τέτοιου είδους ειδήσει σε ευρύτερο κοινό. Καταφέραμε να το εντάξουμε αυτό στον προϋπολογισμό του 2015. Εσείς θα, μπορούσατε να μας διαβεβαίωσετε ότι και το 2016 θα συνεχίσει μια τέτοια χρηματοδότηση. Θα ήθελα να απαντήσω ο Επίτροπος σε αυτό τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαφείς προσδοκίες από τα κράτη-μέλη και από τον προεκλογικό αγώνα και σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Και προτίθεται λοιπόν να βάλει προτεραιότητε στη ε, νομοθεσία, δηλαδή να κάνει πιο λίγα πράγματα και κατά δεύτερον να κοιτάξουμε πού μπορούμε να έχουμε πιο απλά νομοθετήματα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τη σχετική οδηγία, αφενός ελέγχουμε κατά πόσον χρειάζονται και πού χρειάζονται μεταρρυθμίσεις τεχνολογικές λόγω της εξέλιξης της αγοράς, που έχει αλλάξει η αγορά και οι συναλλαγές και κατά δεύτερον θα ελέγξουμε πού είναι τα πράγματα υπερβολικά περίπλοκα, υπερβολικά γραφειοκρατικά. Πού υπάρχουν ενδεχομένως ε, περιθώρια βελτίωσης και απλούστευσης. Αλλά να σας πω ε, ότι σύμφωνα με την δική μου εκτίμηση έως σήμερα πιστεύω ότι χρειάζεται ε, ανανέωση. Αυτό τα μέτρα refit της ε, εκ των υστέρων δηλαδή προσαρμογής, να δούμε πόσο θα, κατά πόσο θα έχουν αποτελέσματα και πολύ γρήγορα στο νέο έτος να προτείνουμε νέα μέτρα. Είχα πολλές επαφές με πολλές, ε, πολλά οπτικοακουστικά κανάλια. την εμπειρία του ΣΔΕΦ Και βλέπουμε λοιπόν ότι στην οδηγία, ε, για την οδηγία αυτή θα πρέπει να προτείνουμε του χρόνου τον Απρίλιο ε, μία πρόταση. Δεν πρέπει να πάρει όμω ε, τρία χρόνια η όλη έγκριση, γιατί στον ψηφοφιακό τομέα οι τεχνολογικέ εξελίξει είναι τόσο μεγάλε και τόσο γρήγορε που θα πρέπει να ισχύουν τα πράγματα αυτά για ένα-ενάμιση χρόνο πριν χρειαστεί η επόμενη αναθεώρηση και ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογικές ε, εξελίξεις και τις νέες εξελίξεις στην αγορά. Στον τομέα αυτό να σας πω ότι θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε επαρκή μέσα στον προπολογισμό προκειμένου τα ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες τεχνολογίε στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών να χρηματοδοτηθούν σωστά με, το, με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς παρόχους ε, τηλεόρασης ε, και ραδιοφώνου από κοινού. Ο ψηφιακός τομέας έως σήμερα δεν αποτέλεσε σημείο επικέντρωσης των διαπραγματεύσεων του TTIP Πιστεύω ότι το θέμα της προστασίας των δεδομένων και το safe harbor του ασφαλούς λιμένα είναι θέματα πιο μεγάλης σημασίας, πιο με υψηλής προτεραιότητας. Αυτό το κοινό κληροδότημα δηλαδή των δεδομένων, αλλά συνολικά η τηλεόραση, οι ταινίε, η εκπαίδευση, οι βιβλιοθήκες δεν πιστεύω ότι αποτελεί, αποτελούν προτεραιότητες των διαπραγματεύσεων, ούτε υπάρχει σχετική εντολή. Και εγώ θα προτιμούσα να σας πω την αλήθεια, ο τομέας αυτό, επειδή δεν περιλαμβάνει μόνο την ε, οικονομία και την αγορά, αλλά αποτελεί και θέμα πολιτισμικό, αποτελεί ένα δημόσιο κληροδότημα, μια δημόσια εντολή. Αν μείνει απαράλλαχτη λοιπόν η ευρωπαϊκή κουλτούρα, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην υποστεί πίεση οικονομική, πίεση της αγοράς, σε ό,τι αφορά θέματα ουδετερότητας του δικτύου. Έχουμε μια ποικιλία ορισμών, προτάσεων ορισμών από διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτάπητος, έχουμε προτάσεις και διατυπώσεις από το Κοινοβούλιο. Το θέμα λοιπόν τώρα ποιο είναι. Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο πριν το Πάσχα θα δώσει στη Λιτωνική Προεδρία τη σχετική εντολή. εκτιμώ και σέβομαι ιδιαίτερα στον Υπουργό και το Υπουργείο του. Τα θέματα αυτά είναι σε καλά χέρια, ε, στα χέρια της Λετωνικής Προεδρίας και εξίσου ικανοί είναι και οι Λουξεμβούργοι που θα ακολουθήσουν. Θα βρούμε λοιπόν διατυπώσεις για την ουδετερότητα του δικτύου που θα αποφύγουν την διακριτική μεταχείριση, που θα διασφαλίσουν ποιότητα και πρότυπα ποιότητας το θέμα λοιπόν είναι ποιε θα είναι οι παρεκκλήσει ε, που θα είναι, δυνατόν, θα είναι δυνατές. Θα μιλάμε μόνο για δημόσια συμφέροντα ή και ειδικέ υπηρεσίε. Εδώ είναι πιο αντιστακτικό, γιατί σε ό,τι αφορά τι δημόσιε καταστροφέ, προστασία από καταστροφέ, δημόσια προστασία, ε, έχουμε όλοι την ίδια από την ίδια άποψη. Για τις ειδικές υπηρεσίες ε, θέλω και είμαι πιο διστακτικός γιατί θέλω να μου πείτε γιατί είναι αυτές οι ειδικές υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Αναφέρατε τα θέματα της Google. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένο. Το θέμα είναι πώς θα πετύχουμε οι πλατφόρμες όπως η Google δεν θα καταργούν τα πνευματικά δικαιώματα. Και τίθεται το θέμα των ε, ημερήσιων εφημερίδων, των περιοδικών. Αύριο, στο μέλλον, θα χρειαστούμε ακόμα, θα χρειαζόμαστε ακόμα εφημερίδες, οικονομικές εφημερίδες, τοπικές εφημερίδες, πολιτισμικές εφημερίδες. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε το περιεχόμενο, όχι όμως το χαρτί, απαραίτητα. Εγώ προτιμώ να διαβάσω εφημερίδα. Ο γιος μου πάλι μόνο στην ταμπλέτα διαβάζει τα θέματα τα αθλητικά. Τις γερμανικές εφημερίδες βέβαια. Στην ταμπλέτα όμως. Αν λοιπόν με τον τρόπο αυτό ε, μειωθεί ο αριθμός ε, των ε, συνδρομητών, γιατί είναι, δεν προτιμούν τις συνδρομές. μείωθεί δραματικά ο ρυθμός των πολυθέντων ε, εντύπων. Και όλα αυτά μεταφερθούν online, τότε πλέον απειλείται η ίδια η ύπαρξη των εφημερίδων. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πρέπει τώρα να δράσουμε. Σε πέντε χρόνια θα είναι πολύ αργά. Θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο είναι δημοσιογράφοι και η εκδοτική οίκη πρέπει να σταθεροποιηθούν και ποιο μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο μέσο και ποιο θα έχει την ε, εξουσία προκειμένου να τηρούνται όλα αυτά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχετική νομοθεσία στη Γερμανία δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ενδεχομένω η Google να αποδεχτεί μόνο μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, μόνο ευρωπαϊκά μέσα. Γιατί αν η Επίτροπος Ανταγωνισμού με επιβάλλει ε, θέματα και μέτρα ανταγωνισμού και ενδεχόμενε κυρώσει, ούτε ίσως αυτό να είναι δυνατόν. Έχετε ε, απόλυτο δίκιο κύριε Αφερχάιεν, οι παιδαγωγοί μας, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι αυτοί που θα λάβουν μία μετέπειτα κατάρτιση. Γιατί σήμερα ένα 14χρονο είναι πιο προηγμένο από τον δάσκαλό του σε θέματα εφαρμογών και ταμπλέτων κτλ. Είναι μεγάλη η συμμετοχή στην καθημερινή ζωή των υπηρεσιών IT, παρόλο που δεν μιλάμε απαραίτητα για υπεύθυνε πληροφορική και αρμόδιε πληροφορική. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολλές θέσεις σπουδών στην πληροφορική Γιατί δεν πρέπει να είμαστε υποδέστεροι από τις άλλες περιοχές του κόσμου σε ό,τι αφορά τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα. Θα πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι και να μην επιτρέψουμε οι άλλοι να είναι καλύτεροι από εμά. Για το Euronet και το Euronews. Για την Euronet και το Euronews. έχουμε τα γλωσσικά σύνορα στην Ευρώπη και γι' αυτό λοιπόν οι υπηρεσίες αυτές κατά κανόνα αποτελούν μία προσφορά της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ένα πρώτο δομικό στοιχείο, αν θέλετε, μιας ευρωπαϊκής δημοσίως γνώμης. Είχα κάνει μια προσφορα της ευρωπης σε παγκοσμιο επιπεδο και ενα πρωτο δομικο στοιχειο αν θελετε μιας ευρωπαικης δημοσίας γνωμης ειχα κανει μια συνεντευξη στη, στη Και αυτό δεν αφορούσε μόνο μία περιφέρεια της Ευρώπης και δεν θα με άκουγαν μόνο σε μία περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά σε πολλές. Και έτσι νομίζω ότι γίνεται μία αποτελεσματική και διασυνοριακή προώθηση και των δικών σας θεσμικών οργάνων. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει τα σχετικά μέσα, και θα επιμένω σε αυτό με την κυρία Γεωργίβα, να ενισχυθούν για να υπάρχει αυτή, αυτά τα διασυνοριακά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Με ρωτήσατε τι γίνεται μεταξύ εμού και του συναδέλφου Ανθιπ, Πώς πάνε οι σχέσεις μας. Πολύ καλά. Γιατί αν υπάρχει ε, πνεύμα ομαδικής συνεργασίας, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Εγώ είμαι αρμόδιος με τις δύο γενικές μου διευθύνσεις, DG Connect για την ευρωπαϊκά ε, θεσμικά ψηφιακά νομοθετήματα και η Γενική Διεύθυνση για την αποθήκευση και την επικοινωνία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η σύνθεση των γενικών διευθύνσεων και ενδεχόμενη βαθμολόγηση είναι δικά μου ζητήματα, δική μου αρμοδιότητα αν αυτό αγγίζει τις αρμοδιότητες και άλλων ε, επιτρόπων, για παράδειγμα τη δικαιοσύνη, την εσωτερική αγορά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θέματα βιομηχανίας, τότε η συντονιστή της διαδικασίας είναι ο συνάδελφος Άνσιπ στις περιπτώσεις αυτές. Συντονιστής μεταξύ των δικών μου προσπαθειών και των εργασιών των άλλων επιτρόπων, προκειμένου να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική και ένα συνεκτικό αποτέλεσμα και να μην ε, γίνεται τελικά να υπάρχουν διαφωνίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αύριο λοιπόν έχουμε δύο συνεδριάσει προ την κατεύθυνση αυτή, όπου ο Άνσιπ θα καλέσει του επιτρόπου που είναι υπεύθυνοι για ψηφιακά ζητήματα, συναρμόδιοι. Εγώ είμαι βασικά ε, υπεύθυνο σε θέματα TSM και copyright και θα συμμετέχουν και οι άλλοι λοιπόν επίτροποι για να αξιολογήσουν καταρχάς τα θέματα copyright από πλευράς νομοθεσίας και από πλευράς οικονομίας της αγοράς και αυτή, αυτός ο συντονισμός θα γίνει από τον Επίτροπο Άντζιπ και μετά αυτά θα επανέλθουν στην γενική μου γενική διεύθυνση. Δεν θα παρεμποδιστεί το δικό μου έργο, αλλά θα ξέρουμε ποιε είναι οι προσδοκίε, ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ των άλλων συναδέλφων τουλάχιστον. Σε θέματα του copyright, πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν έχω κάποια προτιμήση, οδηγία ή κανονισμός. Το θέμα είναι πόσο σε βάθος θέλουμε να περάσουμε. Το θέμα λοιπόν είναι ε, σε τι έυρος θέλουμε να κινηθούμε. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ανοιχτοί, θα πάρουμε οδηγία. Αν θέλουμε πιο δεσμευτικούς κανόνες, να υπάρχουν συγκρίσιμους κανόνες, αυτό σημαίνει ότι θα προτιμήσουμε μάλλον κανονισμό και πιο δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλος δε, σε ό,τι αφορά τις νομικές αρχές, τις ε, ρυθμιστές. Για μια ψηφική αγορά καλύτερα θα ήταν να είχαμε μία αρχή, αλλά ξέρω ότι τα κράτη-μέλη θα ζήσουν πολλά ακόμα σε ό,τι αφορά τον δρόμο του εξευρωπαϊσμού. Αλλά η αρμοδιότητα για τις νομικές αρχές δεν θα δοθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ περιορίζομαι σε έναν καλύτερο συντονισμό. Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς ρυθμιστές λοιπόν, Η ΆΙΖΑ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των ενεργειακών αρχών, είχε πολύ πιο πολλέ αρμοδιότητε σε περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία, για παράδειγμα, για ανάληψη τέτοιων ε, Ε, πρωτοβουλειών σε περίπτωση που υπήρχαν πάνω από 30 για παράδειγμα νομοθέτης. Μία από τις επόμενες οδηγίες θα αφορά τις αρμοδιότητες του, του Μπέρεκ και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δω πόσο ομιλητές έχουμε. Οχτώ ευρωβουλευτές. Σας παρακαλώ να είστε συντομότατοι. Το πολύ 1,5 λεπτό, αλλιώς δεν έχουμε χρόνο. Ο Ζηλό. Και μετά ο κύριο Γραμματικάκης. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είσαστε εξαίρετος. Δύσκολο είναι το σημερινό σας έργο και το κάνετε με μεγάλο ταλέντο. Τρεις ερωτήσει για τα δικαιώματα δημιουργού, έτσι. Για τα γαλλικά μας θέματα βέβαια. Εξηγήσατε ότι υπάρχουν διάφορες οδηγίες και ότι έπρεπε να αναδιατυπώσουμε, εσείς είπατε, ε, αυτές τις οδηγίες και να έχουμε ίσως μία. Αν είχαμε λοιπόν μία οδηγία, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τα δικαιώματα δημιουργού. Θα μπορούσαμε να περάσουμε από τη γαλλική έννοια του γαλλικού δημιουργού στην ε, ευρωπαϊκή έννοια του γαλλικού δημιουργού στην ευρωπαϊκή έννοια για να μπορέσουν και οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, ε, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, εν να λάβουν δίκες ε, απολαβές. Να ξεπεράσουμε τη γαλλική έννοια και να πάμε σε μια ευρωπαϊκή έννοια, λοιπόν. Αυτό για την εδαφικότητα. Δεύτερο θέμα, η μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου. Θα είναι ένα τεράστιο θέμα για την Κομισιόν, αλλά και για το Κοινοβούλιο. Η δυνατότητα μεταφοράς και τρίτον, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, ή μάλλον, εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της οδηγίας του, του κανονισμού για το θέμα της προστασίας της δημιουργικότητας στην Ευρώπη και της προστασίας απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον εμείς ως Κοινοβούλιο και εσείς ως Κομισιόν. Δηλαδή, το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεύτερον το θέμα το νομικό. Γιατί νομικός πώς πρέπει να υπάρχει μία και μόνο ε, νομική δυνατότητα μεταφοράς, ας πούμε. Όχι διάφορες ε, ερμηνείες. Ο κύριος Δραματικάκης. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία του Επιτρόπου εδώ γιατί κάλυψε πάρα πολλά θέματα και κυρίως έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα ασαφές αλλά πάρα πολύ χρήσιμο για μας. Εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων γιατί κύριε Επίτροπε νομίζω ότι η αντίθεση αυτή μεταξύ χριστών και δημιουργών είναι φαινομενική ίσως και πολλές φορές τεχνική διότι κάθε δημιουργός επιδιώκει προφανώς την ευρύτερη δυνατή διάδοση του έργου του. Το κλειδί λοιπόν, το δύσκολο κλειδί, το είπατε ήδη για τη συζήτηση της μεταρρύθμισης, είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων και καθ' όλη την παραγωγική διαδικασία. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τους δημιουργούς, τους κατόχους δικαιωμάτων, τους παρόχους υπηρεσιών, τους εκδότες, τις μηχανές αναζήτησης και άλλους ο νουκάστη αριθμός, όπως λέμε στα αρχαία ελληνικά. Εκεί λίγο θα ήθελα παραπάνω διευκρινήσεις. Πώς σκοπεύετε να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία και κυρίως πώς θα αποσαφινιστεί και θα προσδιοριστεί ο ρόλος των μεσαζόντων. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Il collega eh, Thank you, Chair. Mr. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θέλω να ανατονίσω, όπως είπατε και εσείς, ότι σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που μας ε, έδωσε η Κομισιόν, υπάρχει έλλειψη 700.000 ατόμων στον κλάδο ICT, τεχνολογίας προφορικής δηλαδή, και εξακολουθεί παρά τις προσπάθειες να υπάρχει απόκληση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στον τομέα αυτόν. Τι παραπέρα βήματα θα αναλάβει η Κομισιόν προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκπαίδευση στην πληροφορική. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις ε, απαντήσεις σας. Την τελευταία εβδομάδα, εδώ σε αυτή την Επιτροπή, συζητήσαμε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για τον κινηματογράφο και σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται ότι μόλις το 1,5% των ε, ταινιών του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου έχουν ε, ψηφιοποιηθεί. Τα δικαιώματα λοιπόν χρήσης ε, θα ε, αποκτήσουν πολύ μεγάλη σημασία στο μέλλον. Νομίζω ότι άλλωστε συμφωνούμε όλοι πόσο σημαντική είναι η αρχιοθέτηση των ε, κινηματογραφικών ταινιών και πόσο σημαντική είναι η προβολή αυτής της πολιτικής κληρονομιάς στο ευρωπαϊκό κοινό. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς πιστεύει η Κομισιόν ότι μπορεί να απλοποιηθεί η απόκτηση αυτών των δικαιωμάτων και η εναρμόνιση των δικαιωμάτων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι δεν απαιτούνται μόνο χαμηλές χρεώσεις συναλλαγών, χρειάζεται να υπάρχει και ενιαία αντίληψη για, το, για τη διανομή, την παραγωγή ε, πνευματικού περιεχομένου. Μόλις μας ζητήσετε να σας βάλουμε και στον κατάλογο, έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που μας αγράψατε αυτήν την εικόνα, τη μελλοντική. Όπως ξέρουμε όλοι, το 87% των ε, αιθουσών κινηματογράφου έχουν ήδη ε, μηχανισμό ε, ψηφιακό. Ε, σε κάποιες χώρες όμως, όπως στη Ρουμανία, αλλά και στη Γερμανία, στην Ιταλία, υπάρχουν ακόμα 300 κινηματογράφοι συνολικά που δεν έχουν αποκτήσει τέτοιον εξοπλισμό. Είναι μικροί ανεξάρτητοι κινηματογράφοι σε μικρές χώρες. και που αποτελούν τη μόνη δυνατότητα όμως ε, πρόσβασης ε, σε πολιτιστικό περιεχόμενο για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους Ευρωπαίους για αυτά τα σινεμά ε, το να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν έχουν τα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν έχω να θέσω το εξή ερώτημα. Η Κομισιόν προβλέπει να χρηματοδοτήσει επιπλέον από το πρόγραμμα Media, ας πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία ψηφιοποίησης. Τι μπορούμε να κάνουμε, ούτω ώστε να δώσουμε σε αυτές τις αίθουσες κινηματογράφου το εξοπλισμό που χρειάζεται και για να μην κλείσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραβοβιέσκη. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Σας συγχαίρω για το πρόγραμμά σας που είναι πολύ φιλόδοξο για το 2015. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, κρατάμε την ανάσα μας για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Καταρχάς, ερωτήσεις τώρα. Για την ε, ταχύτητα υιοθέτηση της νομοθεσίας. Η κατάσταση είναι τέτοια που η τεχνολογία είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την νομοθεσία. Πάντα. Παρακολουθείτε το Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο, τα δοηφορικά συστήματα, τα χερσαία. Όλα αυτά είναι προγραμματισμένα μέχρι το 2020. Θα προσπαθήσατε να μειώσετε το τεράστιο άνοιγμα, ανάμεσα, την ψαλίδα αυτή ανάμεσα στην νομοθεσία και στην τεχνολογία. Δεύτερον, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Σαμπίνε Φερχόιγγεν, οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του TTIP είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εσείς τι θα υπερασπιστείτε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, τι εξαιρέσεις, παραδείγματος χάρη, θα προασπίσετε σε αυτές τις διατλαντικές ε, διαπραγματεύσεις. Τρίτον, το κόστος της περιαγωγής για τους νέους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές σας για το 2015. Μέχρι ποιο σημείο είσαστε αισιόδοξο και τι πιστεύετε ότι είναι δυνατό να πετύχουμε ούτω ώστε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος της περιαγωγής. Ε, επίσης, και εγώ σα εύχομαι καλή τύχη για την υλοποίηση αυτών των στόχων που είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Η κυρία Ward. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο και τεχνικό το θέμα αυτό. Το, ερώτημα, το ερώτημά μου είναι φιλοσοφικό, αλλά είναι σοβαρό παρόλα αυτά. Είσαστε ο Επίτροπο της ψηφιακή οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτό το χαρτοφυλάκιο, τι θα ε, ε περιλάμβανε αν οι λέξει είχαν διαφορετική σειρά. Αν ήσασταν ο επίτροπο της Κοινωνίας και της ψηφιακή Οικονομίας, ας πούμε. Ακούω πολλά για αγορέ. το πολιτιστικό τομέα, τους τεχνικούς κανόνες και τους κανονισμούς. Αλλά δεν ακούω και πολλά για τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Πέρα από την κυβερνοασφάλεια ή για το πώς λειτουργούμε ως καταναλωτές. Νομίζω ότι ο, το χαρτοφυλάκιό σας μοιάζει σαν το φτωχό, ας πούμε, συγγενή αυτού που θα θέλαμε. Και στην πραγματικότητα μιλάτε για το πολιτισμό, μιλάτε για το παρελθόν, για την προστασία του, της παρελθούσας πολιτιστικής κληρονομιάς παρά για την δυνατότητα, ας πούμε, ε, δημιουργικότητας. Ε, μπορείτε να δώσετε μια ισορροπία στο χαρτοφυλάκιό σας, ώστε να προωθεί λιγάκι τις φιλοδοξίες της κοινωνίας, να είναι πιο δίκαιο για την κοινωνία, αν θέλετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο κ. Σκουντεύσκη. Γκρασνοντεύσκη, λέει. Διορθώνει η Πρόεδρος, δύσκολη η προφορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δύσκολο το όνομά μου. Ειδικά τα πολωνικά ονόματα εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, όλα τα ονόματα τα, προ, τα σαν ένα. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε λοιπόν εμείς ποιος, όταν αναφέρεται το όνομά του. Είναι πολύ ωραία η γλώσσα μας, ότι είναι δύσκολη, σας ενθαρρύνω να τη μάθετε όλοι. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου, αν μου επιτρέπετε. Θα μπορούσα και εγώ να μιλήσω αγγλικά ή γερμανικά, αλλά όχι, θα μιλήσω πολωνικά. Και τώρα έχω μια ερώτηση. Καταρχάς, μια γενική ερώτηση. Πολύ πρόσφατα τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η Φιλανδία σταμάτησε να μαθαίνει στους μαθητές στα σχολεία πώς να γράφουμε το χέρι. Αποφάσισε δηλαδή να χρησιμοποιούν μόνο το πληκτρολόγιο στη, Φιλανδία. Είναι ένα παράδειγμα μεταξύ πολλών άλλων που μας δείχνει τη σημασία της ε, ανάπτυξης του ίντερνετ. Οποιαδήποτε τεχνολογική πρόοδος είναι καλή φυσικά, αλλά μπορεί να περιορίσει και τις δυνατότητές μας. Και ξέρουμε ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι πάντα θετική για την κουλτούρα. Μπορεί να είναι και επιβλαβής για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Αρκεί να δείτε τι συμβαίνει στα κοινωνικά μέσα, στη, ας πούμε, ο δημόσιος διάλογος στη χώρα μου, επειδή διεξάγεται κυρίως μέσα από αυτά τα κοινωνικά μέσα, ε, έχει φτωχύνει. Εσείς ως αρμόδιος επίτροπος για αυτά τα θέματα, πώς αντιμετωπίζετε την παραδοσιακή πολιτιστική κληρονομιά. Έχω στο μυαλό μου τα βιβλία ας πούμε. Ένα βιβλίο είναι κάτι το οποίο είναι αντικατάστατο. Έχω επίσης στο μυαλό μου μια ομιλία που κάνει κανείς διαζώσεις ένας ας πούμε καθηγητής. Αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει ε, το βιντεάκι ας πούμε που βλέπουμε στις ταμπλέτε ταμπλέτες μας, στις εικόνες. Όλες αυτές τις δεξιότητες πρέπει να τις διατηρήσουμε. Φυσικά οι καθηγητές θα πρέπει να ξέρουν από ίντερνετ, να ξέρουν από τα νέα μέσα ενημέρωσης. Εσείς είσαστε πολύ ενθουσιώδεις σε αυτή την προπαγάνδα. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και η γραφή και η ανάγνωση με την παραδοσιακή έννοια των όρων αυτών είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε κάποιες ε, δυνατότητες, κάποιες ιδιότητες, κάποια προσόντα. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, ας πούμε. Και πρέπει να ενθαρρύνουμε τη Γερμανία και να τη θαυμάσουμε που το κάνει. Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τα όρια αυτής της αγοράς. Δεύτερη ερώτηση, ίσως λιγότερο γενικόλογη. Μιλήσατε για τα δικαιώματα δημιουργού. Εμείς λάβαμε αιτήματα από, διάφορα, από διάφορους κύκλους από διάφορους χώρους που μιλάνε για φόβο αποδυνάμωσης των δικαιωμάτων δημιουργού σε εθνικό επίπεδο. Οι συνομιλητές μας φοβούνται ότι θα υπάρξει μια συγκέντρωση. Θα υπάρξουν μονοπόλια ή ολιγοπόλια, ας πούμε. Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, μπορούν να κυριαρχήσουν την αγορά μας στο σινεμά. μπορεί να υπάρξει μια κυριαρχία της αγοράς και στα βιβλία και στο σινεμά από κάποιους οίκους, από κάποιους ομίλους πάρα πολύ δυνατούς. Αυτό θα μπορούσε να αμφισβητήσει και να υποσκάψει την, ε, τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχετε υπόψη σας όταν εκπονείτε νέες οδηγίες. Αυτό θα να σας ρωτήσω. Ε, Σκέφτεστε αυτές τις αξίες που πρέπει να διατηρήσουμε. Προσέχετε την πολιτιστική πλήρω ε, ποικιλομορφία. Ο κύριος, ο κύριος ε, Διακόνου. Και εγώ έχω λιγάκι, ε, ταυτίζομαι ας πούμε με τον προλαλήσαντα. Φοβάμαι αυτό το ψηφιακό πυρετό που μπορεί να ακυρώσει ορισμένα πράγματα παλιά που υπάρχουν, που είναι ποιοτικά και που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Προηγουμένως, ας πούμε, μιλήσαμε για το βιβλίο, σε υπόθεμα χαρτιού, έτσι. Αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για τεχνολογίες, υπάρχει ένα υπόθεμα, έτσι. Και πάντα μιλάμε για το υπόθεμα και και αγνοούμε το περιεχόμενο. Εμείς αυτό που θέλουμε ένα, είναι ένα ευρωπαϊκό περιεχόμενο ποιοτικό. Στη συνάντησή μας θέλω να μιλήσω για μια παλιά συνάντηση ή μάλλον για μια πρόσφατη συνάντηση που κάναμε ε, στην οποία συμμετείχατε Δηλαδή, θα θυμάστε τι ακροασει για να, γίνετε, επιβεβαιωθείτε ω επίτροπο. Είχα εντυπωσιαστεί τότε από την ε, παρέμβασή σας. Είχατε μιλήσει για την ε, δύναμη του σινεμά, για τη σημασία που είχε η μεγάλη οθόνη, ας πούμε, όταν ήσασταν νέο. Ήταν ο χώρος που μπορούσαμε να συναντήσουμε άλλου ανθρώπου. Είχε μεγάλη σημασία η, η αίθουσα του κινηματογράφου. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον εξυγχρονίσουμε τον κινηματογράφο, το σινεμά δηλαδή την αίθουσα, αλλά χωρίς να χάνουμε τις παλιές αξίες. Το βιβλίο, την λειτουργία του, το, την αίθουσα κινηματογράφου και, την, και το ρόλο της, την εφημερίδα που διαβάζετε κάθε πρωί κτλ. κτλ. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό που ονομάζουμε Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ταινίας. Κάτι τη γνώμη μου μοιάζει με μία άσπρη Δεν ξέρουμε και πολλά. Δεν ξέρουμε πότε θα πεταχτεί από το νερό και τη στιγμή που θα πεταχτεί με τι μοιάζει. Τέλο πάντων, το ερώτημά μου είναι το εξή. Πώ και πότε μπορούμε να δούμε αυτή την άσπρη φάλαινα. Δηλαδή αυτό το φόρουμ του Ευρωπαϊκού Φιλμ που ακόμα δεν το έχουμε δει. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ε, διατυπώθηκαν. Έχετε 20 λεπτά για να απαντήσετε. Περίπου. Είμαι πεπισμένος ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος μπορεί να έχει μέλλον και ότι στον τομέα αυτό πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να βελτιστοποιήσουμε την στρατηγική μας σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ε, και ο κλιματογράφος αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά μας. Χρειάζεται η χρηματοδότηση του κινηματογράφου σε εθνικά, στα κράτη-μέλη. Ε, χρειαζόμαστε επίσης κρατικές ραδιοφωνίες δημόσιες ραδιοφωνίες που επιδοτούνται από το κράτος δηλαδή και δεν λειτουργούν μόνο με ε, έσοδα από διαφημίσεις και ε, τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες αποδεχτήκαμε αυτό το καθεστώς. Αυτή η δυτή λοιπόν ε, κατάσταση λέγαμε ότι εξασφαλίζει την ποιότητα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν και οι δημόσιοι φορείς ραδιοφωνίας να δουν και να αντιληφθούν τον ρόλο τους με αυτόν τον τρόπο και να μην προσπαθεί απλά να αποσπάσει μερίδια ακροαματικότητας, θεαματικότητας από τους ιδιωτικούς σταθμούς. Αλλά να προσέξει και το, την ε, πολιτιστική, την ποιοτική διάσταση. Υπάρχουν και κίνδυνοι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να, υπα... να απαγορεύσουμε την τεχνολογία. Μπορούμε όμως να θέσουμε συγκεκριμένου κανόνες. Πριν από 8 χρόνια δεν υπήρχαν iPhone στην αγορά. Και πάω στοίχημα ότι η τεχνολογική επανάσταση θα επιταχυνθεί. Τα επόμενα πέντε χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας, των εφαρμογών, του software και του hardware θα έχει θα είναι τόσοι όσοι υπήρξε τα τελευταία 10 χρόνια. Αν πάτε στα ερευνητικά εργαστήρια, αν μιλήσετε με ανθρώπους από τις startup εταιρείες, θα διαπιστώσετε ότι τα πάντα κινούνται με τεράστιες ταχύτητες, με φοβερή δημιουργικότητα. Και φυσικά υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, αυτό που αποτελεί το καύσιμο δηλαδή αυτής της ε, τεχνολογικής πρόοδου. Καθήκον δικό, μας, καθήκον δικό μας είναι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο, το ρυθμιστικό. Στους εφήβους για παράδειγμα πρέπει να μιλήσουμε, στο θέμα των εφήβων πρέπει να μιλήσουμε για παράδειγμα για την προστασία της συγκεκριμένη ε, πληθυσμιακής ομάδας για να δυσκολέψουμε την πρόσβαση στην πορνογραφία, σε περιεχόμενο που εξοραίζει τη βία, σε περιεχόμενο που εξοραίζει εγκλήματα. Γι' αυτό και όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οπτικοακουστικής οδηγίας. Δεν ανοσυχώ τόσο πολύ για το διάβασμα στο τάμπλετ, όσο για την γραφή πρέπει να σας πω. Τώρα, το αν διαβάζει κανείς ε, ένα κείμενο σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή δεν έχει ε, μεγάλη διαφορά. Είναι όμως σαφές ότι το να γράφει κανείς μπορεί τελικά να αμφισβητηθεί ως ε, ικανότητα των ανθρώπων. Και αποτελεί πολιτισμικό αγαθό η ικανότητα να γράφει κανείς. Γιατί όταν είσαι υποχρεωμένος να γράψεις, σκέφτεσαι και περισσότερο και πιο σε βάθος αυτό που πας να γράψεις. Ενώ αντίθετα αν γράφεις κάτι στο τάμπλετ, γράφεις αρκτικόλεξα, συντομογραφίες, διάφορα σημεία στήξης. Μπορεί να ακούγομαι συντηρητικός, αλλά εγώ θέλω τουλάχιστον για την επόμενη γενιά μαθητών να διατηρηθεί η διδασκαλία της γραφής ως σημαντικής ικανότητας για τους νέους. Δεν πρέπει να, να παραιτηθούμε από αυτό. Μπορεί σε 20 χρόνια να μην χρειάζεται πλέον να γράφουν οι άνθρωποι. αυτό, ένα, αυτό μπορεί να, να ισχύει. Αλλά είναι σημαντικό να γράφει κανείς και να μπορεί να γράφει και στο χώρο εργασίας τους και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να εγκαταλείψουν βεβαιασμένα τη διδασκαλία της ε, ε, γραφής. Ναι, σκοπός μου είναι η θέσπιση ευρωπαϊκού δικαιώματος δημιουργού. Να σας πω, αν κάποιος μουσικός στην ε, περιοχή μου ε, γράψει ένα τραγούδι για την ομορφιά των Άλπων, αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να πουληθεί ποτέ στη Ρήγα ή στη Λισαβόνα. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι όταν ένα πολιτιστικό περιεχόμενο έχει τοπική διάσταση μπορεί κανείς να πει ότι εδώ υπερισχύει η αρχή της ε, επικουρικότητας. Εδώ δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε ε, ευρωπαϊκούς κανόνες αξιοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων κτλ. κτλ. Θα περιοριστούμε δηλαδή με άλλα λόγια σε έργα που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Είναι αλήθεια ότι μπορείτε σήμερα πια να κατεβάσετε όποιο τραγούδι θέλετε και να μην πληρώσετε τίποτα. Παλιά υπήρχαν οι δίσκοι βινιλίου και πουλιούνταν αυτοί οι δίσκοι σε καταστήματα. Όταν κάποιος αντέγραφε τη μουσική από δίσκο σε κασέτα, ήταν παράνομο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, εξακολουθούσε για πολλά χρόνια να υπάρχει ένα προϊόν το οποίο πολιόταν στα καταστήματα. Και, από, και με αυτόν τον τρόπο ο δημιουργός είχε εισόδημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο και για το μέλλον. Αν ναι, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε από τα YouTube, τα Google κτλ. κτλ να ζητούν κάποιο ποσό από κάθε έναν που κατεβάζει μουσική και αυτό το ποσό να το μεταβιβάζουν στο δημιουργό. Αυτό είναι το αποφασιστική σημασία σημείο. Αν δεν καταφέρουμε να χαράξουμε ένα τέτοιο δρόμο, δεν θα υπάρξει άλλη γενιά δημιουργών. Αν δεν υπάρχουν αξίες, αν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο. Καταλάβατε γιατί ελάχιστοι είναι απλώς αλτροιστές. Οι περισσότεροι δημιουργοί κάνουν τη δουλειά που κάνουν για να κάνουν και καριέρα και για να μπορέσουν να θρέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Θέλουμε λοιπόν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών να συζητήσουμε την αύξηση των ε, θέσεων κατάρτισης στην πληροφορική. Να διαπιστώσουμε δηλαδή ποιες θα είναι οι ανάγκες μας το 2020, 2025, 2030. Ποια είναι τα καλύτερα, ποια είναι τα χειρότερα σενάρια, πόσους χρειαζόμαστε τελικά, πληροφορικάριους δηλαδή. Και στη συνέχεια θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένα μέτρα έως ότου η Ευρώπη καταφέρει να πετύχει τον αριθμό ειδικών στην πληροφορική που χρειάζονται και ενδεχομένως να προσελκύσουμε και ανθρώπους από την Ινδία, ώστε να μην πηγαίνουν στην ΣΥΠΑ, αλλά να έρχονται σε μας Οι Ινδοί δεν έρχονται εδώ στην Ευρώπη γιατί δεν υπάρχει ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν 28 διαφορετικές αγορές που θα πρέπει να το αναδιοδοτήσουν η κάθε μία ξεχωριστά. Όταν λοιπόν υπάρχουν 28 αγορές με διαφορετικούς κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κτλ. κτλ. Το γραφειοκρατικό βάρος είναι υπερβολικό για να έρθει κανείς εδώ. Γι' αυτό και οι startups πηγαίνουν στην Αμερική 330 εκατομμύρια καταναλωτές και ένα σύνολο κανόνων. Γι' αυτό είναι ουσιώδης η σημασία της δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ε, αναφερθήκατε και στο θέμα της ε, ταχύτητας, ότι αργήσαμε. Ισχύει. Γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε τον φιλόδοξο στόχο, να μην καθόμαστε να συζητάμε τώρα για τρία χρόνια, αλλά να προχωρήσουμε γρήγορα. Όχι όπω έγινε με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που χρειαστήκαμε 3,5 χρόνια από τη στιγμή που η Vivian Redding υπέβαλε την πρότασή τη. Γιατί? Γιατί τα κράτη-μέλη δεν ήταν πεπισμένα για τι τις αρχέ τη πρόταση. Εμεί πρέπει τώρα να αξιοποιήσουμε την ε, δυναμική που έχει δημιουργηθεί και να ρωτήσουμε, συνάδελφοι, είστε πρόθυμοι, είστε έτοιμοι να συμβάλλετε στην ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Ναι ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι οι υπουργοί των εθνικών κυβερνήσεων θα πρέπει να ασχοληθούν και με τα καθήκοντά τους στο Συμβούλιο. Αν γίνει κατανοητό αυτό, τότε θα προχωρήσουμε και θα, θα έχουμε κερδίσει. Και νομίζω ότι το θέμα της ψηφιακής στρατηγικής είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αλλιώς οι διάφορες Google δεν θα έχουν κανένα σεβασμό στον κατακαιρματισμένο, στην κατακαιρματισμένη ε, αγορά μας. Για το TTIP. Ο τομέας αυτός ε, που σας ενδιαφέρει εμάς, οι ταινίε, τα μέσα, η εκπαίδευση, ο ηλεκτρονικός πολιτισμός, οι ε, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, δεν αποτελούν ε, καθόλου αντικείμενο διαπραγματεύσεων, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο μια αγορά που έχει να κάνει με θέμα βασικής προμήθειας, βασικών συμφερόντων, μόρφωσης, κουλτούρας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μείνουν έξω αυτά και η εντολή που έχει δοθεί ω τώρα δεν έχει θέσει τέτοιε προτεραιότητε για την δομή διαπραγμάτευση της συμφωνία TTIP για το roaming, την περιαγωγή. Η έκθεση Berg του Δεκεμβρίου έκανε μια έξυπνη ανάλυση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η περιαγωγή είναι απαραίτητη. Σε μια ενιαία αγορά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διασυνοριακοί δασμοί. Αν σήμερα στη Γερμανία πάει κανείς από το Άχεν και τηλεφωνήσει 500 ε, χιλιόμετρα ε, απόσταση μέσα στη Γερμανία ή τηλεφωνήσει 30 χιλιόμετρα απόσταση στο Βέλγιο, γίνεται το εξή περίεργο στα 30 χιλιόμετρα απόσταση, επειδή είναι διασυνοριακή η κλίση, είναι πιο ακριβό τηλεφώνημα από ό,τι στην πρώτη περίπτωση. Αυτό είναι παράλογο λοιπόν. Τα εθνικά σύνορά μας ε, προέρχονται από την εποχή του Ναπολέοντα, από το συνέδριο τη Βιέννης, από τη διάσκεψη τη Βαρσαλιών και από τη Γιάλτα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ο Ναπολέοντας δεν είχε φανταστεί ακριβώς έτσι την ψηφιακή επικοινωνία. Υπήρχε τότε το περιστέρι. Γι' αυτό λοιπόν τα εθνικά σύνορα δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τα ψηφιακά μας συμφέροντα, με τα ψηφιακά μας δικαιώματα και τις ανάγκες μας η έννοια ψηφιακή οικονομία και ψηφιακή κοινωνία ήταν δική μου ιδέα και το έθεσα αυτό σκόπιμα γιατί στην ψηφιακή σελίδα πιστεύω ότι υπάρχει και οικονομικός παράγοντας αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις. Πολλές κοινωνικές ευκαιρίες, κοινωνική κίνδυνοι και προκλήσεις. Άρα δεν είναι μόνο τεχνολογική η επανάσταση αλλά μεγάλη πρόκληση για την κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να επισημαίνουμε τους, τους κινδύνους. Δεν θα πρέπει όλα να μπαίνουν στο δίκτυο. Να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία του Twitter, του WhatsApp, γιατί μιλάμε και πάντα για προστασία προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη κύριε Μόρντεν ξεχάσαμε να σας δώσουμε το λόγο. Ε, θα σας το δώσω ως τελευταίο ομιλητή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Άκουσα αυτό που μας είπατε διάφορες φορές κατά τη διάρκεια της παρέμβασής σας για τη δυνατότητα επιτάχυνσης για της οδηγίας για το οπτικό ακουστικό και το θέμα της μεταρρύθμισης του copyright και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ούτως ή άλλως ε, επιταχύνονται τα πάντα στο, στο ψηφιακό χώρο, επομένως οποιαδήποτε νομοθέτημα για αυτά ε, καθίσατε γρήγορα απαρχαιωμένο. Τώρα, για το TTIP με το οποίο σχολείστε, θα υπάρξει επιτάχυνση αυτής της ε, οδηγίας ή μεταρρύθμιση της οδηγίας, δεδομένων αυτών των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, πώς κολλάνε τα δύο θέματα. Από τη μία οδηγία, από την άλλη η Δεν θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθούμε σε δυσκολία επειδή θα είμαστε ακόμα έτοιμοι ή, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουν ε, οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό ακριβώς παίρνω τον λόγο. Γιατί δεν θα είμαστε πάλι έτοιμοι. Ξέρετε πολύ καλά τι πρόβλημα έχει η ανεργία στον δημιουργικό χώρο, στον κλάδο αυτό. Θα ήθελα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια Ευρωπαίων που δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο και σε επίπεδο ΑΕΠ έχει σημαντικό βάρος ο ε, οπτικοακουστικός χώρος ε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορείτε να απαντήσετε, Επίτροπε. Οι γρήγορε διαπραγματεύσει ε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και τσαπατσούλικε. Ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προέρχεται από το 2012. Τα δύο πρώτα χρόνια κοιτάξαμε πολύ λιγότερα από το τελευταίο εξάμεινο. Σε μισό χρόνο δηλαδή το Συμβούλιο κατάφερε πιο πολλά από τα δύο πρώτα χρόνια. Στο θέμα TSM, για την οδηγία δηλαδή για την ενιαία ε, αγορά για τις τηλεπικοινωνικίες, για την περιαγωγή, για την ουδετερότητα του δικτύου, αποφασίσω την άποψή σας το 2013. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είχε τόσο σχετική εντολή δεν ε, είναι Καλό. Δεν είναι εντάξει. Τόσο καιρό μετά. Πρόκειται για μια καθυστέρηση την οποία δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και να επιτρέψουμε πλέον. Αν είχαμε το Σεπτέμβριο εντολή του Συμβουλίου, θα μπορούσαμε να βρούμε γραμμέ σεμιβασμού για το ρόμι, για την περιεγωγή και για την ουδετερότητα του δικτύου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και εσεί είσαστε εξαγριωμένοι και θυμωμένοι. Άρα θέλω να εργαστούμε εντελεχώς, αλλά και γρήγορα για τα οπτικοακουστικά, για παράδειγμα. Θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για το ReFit του 2015 και του χρόνου θα κάνω την πρότασή μου για την μεταρρύθμιση, για την ανανέωση, τα νέα περιεχόμενα σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές ε, εξελίξεις, καλό θα ήταν το συντομότερο δυνατόν να συμφωνήσουμε. Όχι σε δύο χρόνια. Τέλη του 2016, αρχές του 2017 θέλω να έχει νομική ισχύ καινούργια οδηγία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια σας. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Να σας πω ότι εκτιμούμε πάρα πολύ και την ε, επιβεβαίωση της ε, πολιτικής εξαίρεσης ε, στα TTIP και θα θέλαμε να δούμε και τι, τι βαθμό, σε ποιο βαθμό και μέχρι που πάει αυτή η εξαίρεση. Στις 7 Φεβρουαρίου είναι η μέρα για, την, για το ασφαλέστερο ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα σε σχέση με τα παιδιά. Πιστεύουμε ότι για τα θέματα του ίντερνετ θα προχωρήσετε. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε και καλή δουλειά, καλή συνέχεια.